Η κυρία Μογκερίνη έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους αγαπητούς μας φίλους. Ε, είναι απόδειξη ότι το έργο που κάνουμε μερικές φορές ε, αφανώς ε, και διακριτικά έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που είστε εδώ. Θα ήθελα να σχολιάσω δύο κυρίως από τα σημεία που επισημάνατε. Βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει κτήμα του αυτή την παγκόσμια στρατηγική και χαίρομαι ιδιαίτερω γι' αυτό γιατί βλέπω ότι μπορώ να υπολογίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί όπω είπατε είναι συλλογική προσπάθεια, συλλογικό το έργο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και συλλογικά μία παρακολούθηση για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα και να το δώσουμε σάρκα και οστά. Μερικοί από εσά ρώτησαν αν τονίζουμε καλύτερα τις αξίες και τα συμφέροντα ή αν τα θεωρούμε σημαντικό στοιχείο των μελλοντικών μας δράσεων, τις αξίες και τα συμφέροντά μας. Η βάση της στρατηγικής και η σαφής ένδειξη της στρατηγικής είναι ότι οι αξίες μας και τα συμφέροντά μας συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ένα στοιχείο των αξιών μας που υπογραμμίζει στρατηγική. Δηλαδή, για να είναι συνεκτική και συνεπής η δράση μας θα πρέπει να διέπεται από τις αξίες μας. Θα πρέπει ε, να τιμούμε τις αξίες μας και στη συμπεριφορά μας και στις πολιτικές μας. Θα επισήμαναν αυτό κάποιοι ευρωβουλευτές. Οποιαδήποτε παγκόσμια στρατηγική ξεκινάει ε, στον οίκο μας και εξαρτάται από την εσωτερική μας δύναμη. Γι' αυτό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό να αναλάβουμε τις κοινέ μας ευθύνες απέναντι στους πολίτες μας αλλά και προς τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, επαναλαμβάνω, συμπίπτουν οι αξίες και τα συμφέροντα που έχουμε. Σκεφτείτε την ανθεκτικότητα, την ανάγκη ανθεκτικότητας που βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Η ανθεκτικότητα των κοινωνιών ε, γύρω μας είναι επένδυση και στη δική μας ασφάλεια. Και όταν αναφέρομαι σε ανθεκτικότητα των κοινωνιών ε, στη στρατηγική, δεν ε, αναφέρω με μόνο στην ισχύ των θεσμικών οργάνων αλλά στην ίδια την αφεκτικότητα των κοινωνιών δηλαδή ε, στους ε, ακτιβιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων στην κοινωνία των πολιτών στη δική τους αφεκτικότητα και στη θέση κάθε πολίτη στην κοινωνία του. Αυτό ανταποκρίνεται μόνο στις αξίες μας, όχι ανταποκρίνεται και στα συμφέροντά μας. Και νομίζω ότι είναι κοινή αυτή η ένδειξη. Και στην περίπτωση αυτή, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η τήρηση και ο σεβασμός των αξιών μας εξυπηρετεί και τα συμφέροντά μας. Και νομίζω θα ήταν λάθος αν θεωρήσουμε ότι είναι αντιφατικά τα συμφέροντα από τις αξίες μας ή αντικρουόμενα. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που επισημάνατε μερικοί. Κάποιοι το έθεσαν αρνητικά και κάποιοι υποθετική σκοπιά, ο κύριος Ντανζάν για το Train and Keep, για την δημιουργία ικανοτήτων στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη και άμυνα. Χρειάστηκε μία τριετία για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε το πακέτο για τη δημιουργία ικανοτήτων στην ασφάλεια και την ανάπτυξη. Και θα σας το πω ξεκάθαρα και σαφέστατα ότι σε καμία περίπτωση δεν αποκλίνουμε ε, από τα αναπτυξιακά μας ε, τους αναπτυξιακούς μας μηχανισμούς και δεν εκτρεπόμαστε προς μια ε, προοπτική ασφάλειας. Όχι. Αλλά όπως λέει και η κοινωνία των πολιτών, σε όποια περιοχή και βρισκόμαστε, στο Σαχέρι, στην Ιγυρία, στο κέρα της Αφρικής, αν σε μια περιοχή ε, δεν ε, υπάρχουν στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας για τον πληθυσμό, ό,τι αναπτυξιακές δράσεις και να αναπτύξετε, είτε δεν θα φτάσουν στους αποδέκτες, είτε δεν θα είναι αποτελεσματικές. Πρώτα θα πρέπει να εξασφαλιστεί το θεμελιώδες δικαίωμα στην ασφάλεια που είναι αλληλένδετο με την ανάπτυξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, μεταφέρουμε πόρους από την ανάπτυξη στην ασφάλεια. Όχι, απλώς λέμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και να αξιοποιούμε τους πόρους μας με συνεκτικό τρόπο και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πληθυσμών. Πάντως ε, αυτό μας λένε όλοι οι συνεργάτες μας ε, και αυτό το χαρακτήρα έχουν όλα τα μηνύματα που λαμβάνουμε, ότι θα πρέπει να εργαστούμε και για την ασφάλεια, όπως συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και την ανάπτυξη. Γιατί δεν νοείται ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη και τα ανάπαλη. Θα πρέπει τώρα να το μεταφέρουμε και στην πράξη. Είναι αλληλένδετα και τα δύο και το χθεσινό πακέτο που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και θα συμβάλλει στην ικανότητά μας να εφαρμόσουμε και τη συγκεκριμένη στρατηγική, την παγκόσμια στρατηγική, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μας που καλύπτουν διαφορετικούς ε, τομεί, αλλά να τα αξιοποιούμε με ολοκληρωμένο και τρόπο συνεργασίας και συνεκτικό τρόπο. Ε, ένα τμήμα της στρατηγικής προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να, μπορούν να, κληθούν να συμμετάσχουν σε διάφορες πτυχές της πολιτικής. Είναι ένα τμήμα τη στρατηγική ε, που το επεξεργαστήκαμε με, με ιδιαίτερη προσοχή όπω θα φαντάζεσαι και ανταποκρίνεται στο γεγονό ότι αφενό πρέπει να διασφαλίσουμε την ενότητα όχι μόνο των 28 χωρών μελών αλλά και των διαφόρων θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό κάνουμε στο πλαίσιο των κοινών θεσμών αλλά σε μερικές περιπτώσεις ε, ίσως ε, επιθυμούμε ή χρειαζόμαστε ή θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε μία χώρα ή μία ομάδα χωρών ή γιατί όχι και κάποιες κοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείες να συμπληρώσουν το έργο που κάνουμε όλοι από εκείνο το συλλογικό μας έργο. Ίσως εκεί έχουμε επιπλέον προστιθέμενη αξία. Το σημαντικό πάντως είναι όλα αυτά να γίνονται με συντονισμένο τρόπο, με σαφή και διαφανή ε, σχέση με τις κοινέ ε, αποφάσεις και στα στα κοινά μας όργανα. Δεν θα με φόβιζαν πρωτοβουλίες είτε κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών, είτε ομάδας ε, κρατών, είτε και ομάδας επιτρόπων. Το βασικό είναι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις να εντάσσονται σε ένα κοινό πλαίσιο και να αποβλέπουν σε ένα κοινό στόχο. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε την προστιθέμενη αξία μας, ακόμη και όταν είναι μερική. Το βασικό είναι να ανήκει σε μια ε, συνεπή, συντονισμένη και συνεκτική πολιτική. Και τώρα έρχομαι στη βασική μας, στην πρωταρχική μας ανάγκη. Το αναφέρατε πολύ από εσά. Η πρωταρχική μας ανάγκη τώρα είναι να ε, διασφαλίσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και να εγγυηθούμε την ασφάλειά τους κάτι τέτοιο απαιτεί δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μία πρόταση που, που κάνατε δεν πρόκειται να την ακολουθήσω. Κάποιος είπε ότι δεν αναφέρεται στα αγγλικά η ανάγκη να ληφθεί περισσότερη υπόψη ε, να ληφθούν περισσότερο υπόψη κάποιες ε, σκέψεις, κάποιες απόψεις που είναι κατά της κοινή ε, ε, προσπάθειας ή της συνεργασίας ε, και κάποιες να γίνουν σεβαστές και φορές που λένε ότι δεν είναι σωστός ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμε πολύ, αλλά δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Αν υπάρχει ένας τομέας όπου είναι αυταπόδεικτο ότι η ασφάλειά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί κοινή δράση, είναι ακριβώς αυτός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τομέας στις εξωτερικές μας δράσεις όπου μία μόνο χώρα από μόνη της, όσο δυνατή και αν είναι, όσο μεγάλη και αν είναι, όσο εύπορη και αν είναι, είναι μόνη της πιο αποτελεσματική από το σύνολο των κρατών μελών. Είτε μιλάμε για την τρομοκρατία, είτε μιλούμε για το εμπόριο, είτε μιλούμε για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Καμία χώρα από μόνη της, όσο ισχυρή και είναι, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Σίγουρα είμαστε ισχυρότεροι ενωμένοι παρά ο καθένας ξεχωριστά. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην ασφάλεια, γιατί οι απειλέ και οι ευκαιρίες είναι παγκόσμιες. Και όλες οι χώρες μας σε σύγκριση με τις υπόλοιπε χώρες του κόσμου είναι μικρές. Ακόμη και οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε παγκόσμιο ε, επίπεδο είναι μικρές. Δεν βρισκόμαστε στην εποχή των αυτοκρατοριών. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτή την πραγματικότητα. Αυτό το βλέπουν οι εταίροι μας και αναγνωρίζουν την ισχύ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή την ισχύ μερικές φορές εμείς δεν τη βλέπουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από την κατάθλιψη που μας χαρακτηρίζει και να αξιοποιήσουμε την ισχύ μας. Γιατί μπορεί κανείς να είναι δυνατός, αλλά αν δεν γνωρίζει τη ρόμη που έχει μέσα του, δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Και όπως είπατε κάποιοι, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική ώστε να μετατρέψουμε το κοινό μας όραμα σε κοινή δράση και να γίνουμε ένας παγκόσμιος εταίρος με αυτοπεποίθηση. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Μερικοί είπατε ότι η στρατηγική παρά είναι φιλόδοξη, ότι είναι ουτοπική, άλλοι είπαν ότι παρά είναι ρεαλιστική αλλά δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Χρειαζόμαστε και, φιλο... και ρεαλισμό αλλά και φιλοδοξία και μία αποστολή. Γιατί βλέπετε πόσο ραγδαία μεταβάλλονται τα πράγματα και εσωτερικά και εξωτερικά. Ε, με τρόπο που πριν από μερικούς μήνες και χρόνια ήταν αδιανόητο. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδρούμε και στις αλλαγές που γίνονται αλλού ή αν έχουμε αρκετή αυτοπεποίθηση να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε τις αλλαγές που γίνονται γύρω μας. Και πιστεύω ότι έχουμε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μας και όλη την δύναμη αρκεί να έχουμε και την πολιτική βούληση να το κάνουμε όπως ε, θέλουν οι πολίτες από εμά έχουν και συμφέρον άλλωστε. Ευχαριστώ. Να περάσω στο επόμενο σημείο, αλλά θα το πει ο πρόεδρος.